Καλημέρα συνάδελφοι, θα αρχίσουμε. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση σχετικά με την επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στην Κύπρο. Τέλη Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα ο κύριος Σταυρακάκης που προείδρευσε τις αποστολή αυτής να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριος σκοπός της αντιπροσωπείας μας ε, της Επιτροπής ήταν ε, ε, η εξέταση της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στο νησί είχαμε μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες και χρήσιμες συναντήσεις. Ε, την πρώτη μέρα στις 26 Σεπτεμβρίου ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο μας παρήχε μια σύντομη ενημέρωση για την επίσκεψη και για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της Κύπρου. Την επόμενη μέρα συναντηθήκαμε με τον Κύπριο Υφυπουργό Αρμόδιο για Ευρωπαϊκά Θέματα, τον κύριο Ανδρέα Μαυρογιάννη, καθώς και με προσώπους της Διαχειριστικής Αρχής για τα διαθροτικά ταμεία και συζητήσαμε διεξοδικά τις εξελίξεις της διαπραγματεύσης για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς και τη νομοθετική δέσμη για τη μελλοντική πολιτική συνοχής μετά το 2013 και τις θέσεις της Κυπριακής Προεδρίας επί αυτών των θεμάτων. Στη συνέχεια είχαμε μια πολύ επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με την Υπουργό Εργασία και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρία Σωτηρούλα Καραλάμπους σχετικά με την τρέχουσα εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, όπως επίσης και για τον μελλοντικό κανονισμό του. Οι συναντήσεις μας με τα μέλη της Κυπριακής Κυβέρνησης ολοκληρώθηκαν με τη συνάντηση που είχαμε με την Υπουργό Εσωτερικών κυρία Ελένη Μαύρου, η οποία μας παρήχε πληροφορίες για τις υποδομές της χώρας, την κατάσταση των δημόσιων μεταφορών, την αστική και αγροτική ανασυγκρότηση και την διαχείριση διαφόρων τύπων αποβλήτων. Συναντηθήκαμε επίσης με τον Δήμαρχο της Λευκοσίας, όπου συζητήθηκε το ζήτημα της διαίρεσης της πόλης και το πώς αυτή επηρεάζει τους ανθρώπους και στις δύο πλευρές της πράσινης γραμμής, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής θα μπορούσε να συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης. Επί του παρόντος, τα δύο μέρη προσπαθούν να ανακτήσουν κάποια κτίρια στην νεκρή ζώνη, προκειμένου να φιλοξενήσουν και να αναπτύξουν πολιτιστικέ δραστηριότητε για να φέρουν πιο κοντά τι δύο κοινότητε. Επίση, με τον Δήμαρχο τη Λεμεσού ανταλλάξαμε απόψει για τη συμβολή τη πολιτική συνοχή στην αναδιαμόρφωση ανάπλαση τη πόλη. Το πρόγραμμά μα περιλάμβανε επίση επιτόπιε επισκέψεις σε μία σειρά από χρηματοδοτούμενα, συγχρηματοδοτούμενα από τα διαφορετικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχή Έργα, οι οποίες μας έδωσαν την ευκαιρία να διαπιστώσουμε από πρώτο χέρι τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται στην πράξη η πολιτική συνοχή. Την τελευταία ημέρα της επίσκεψής μας συναντηθήκαμε με μέλη των Επιτροπών Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εσωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με την ανάγκη για σύγκληση μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωση, καθώς και για ένα βιώσιμο μέλλον για τις γενιές του αύριο. Συνολικά η επίσκεψη αυτή έδωσε την ευκαιρία στα μέλη της αντιπροσωπείας μας να ανταλλάξουν ιδέες με τους εκπροσώπους των περιφερειακών και τοπικών αρχών και να αξιολογήσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των διαθροτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής στη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές της. Επίσης, αξιολογήθηκε ο τρόπος με τον οποίο έχει υλοποιηθεί η πολιτική συνοχή για την προώθηση της επανένωσης του νησιού. Επιπλέον, συζητήσαμε ει βάθο τι γραμμέ που υπερασπίζεται η Κυπριακή Προεδρία κατά τη διάρκεια των τρεχουσών διαπραγματεύσεων και εκφράσαμε τι ανησυχίε τη Επιτροπή μα, καθώ και τη θέση τη αναφορικά με την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι στόχοι που τέθηκαν για την επίσκεψή μας επιτεύχθηκαν στο σύνολό τους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αυτά είχα να παρουσιάσω και αν κάποιος συνάδελφος από την Επιτροπή θέλει να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο. Υπενθυμίζω επίσης στους συναδέλφους ότι ο Γιώργος προείδρευσε τη αντιπροσωπείας και η Κωνσταντζα Κρέλ ήταν εκεί και ο κ. Φανίστερα, ο Νικολάτσικ, Πετρουγιώχαν, Καμάνεν στην αντιπροσωπεία αυτή. Οπότε αν έχει κάποιος, σας, κάποιος από εσά να προσθέσει κάτι, τώρα είναι η στιγμή. Ερωτήσεις? Όχι από ό,τι βλέπω, ούτε σχόλια. Καλώ δεν χρειάζεται έτσι καλώ να πάρουμε καμία απόφαση από αυτού. Την έκθεση θα τη στείλω και στη διάσκεψη των Προέδρων, γιατί έτσι καλώ πρέπει να του ενημερώνουμε για τα ταξίδια μας. Ευχαριστούμε Γιώργο και πάλι. Τώρα σας ενημερώνω για τις αποφάσεις που λήφθησαν ε, από τους συντονιστές ε, των πολιτικών ομάδων χθες. Πρέπει να επικοινωθούν από την Επιτροπή μας χθες Λοιπόν, αποφασίσαμε για το ποιος θα πάρει την κάθε έκθεση. Όσον αφορά τα ταμεία για την ευρωπαϊκή ενίσχυση στους πιο αδύναμους, την ανέλαβε η Γκουε. Την έκθεση για την οδηγία για την πρόθεση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ανέλαβε η Άλντε. Τις γνωμοδοτήσεις τώρα. Γνωμοδότηση για την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού για την απαλλαγή 2011 την ε, πήρε το ΕΛΚ. Ο σχεδιασμός πολιτικής ε, lock and trends με δημοσιονομικές επιπτώσεις την πήρε η Το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου το πήρε το ΕΛΚ. Για την κοινωνική στέγαση οι σοσιαλιστές. Οίκο ε, καινοτομία ανάπτυξη οι σοσιαλιστές καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη την πήρε η Άλντε, πρόθεση ευρωπαϊκής στρατηγικής και τεχνολογίας για τις μεταφορές την πήραν πράσινη, εφαρμογή της στρατηγικής για την νεότητα, η ΓΚΟΕ. Ζητούμε από τους πολιτικούς συντονιστές να ενημερώσουν την γραμματεία σήμερα, μέχρι το τέλος της ημέρας, για το όνομα του εισηγητή, του συντάκτη γνωμοδότησης. Πρέπει επίσης να συζητήσουμε και τις μελλοντικέ μας εκθέσεις, ιδίας πρωτοβουλίας για το 2013. Είναι κάτι που το συζητήσαμε χτες και αποφασίσαμε ότι το Δεκέμβριο στη συνεδρίασή μας θα πρέπει τελικά να αποφασίσουμε για αυτά τα θέματα. Στο μεταξύ δηλαδή οι πολιτικές ομάδες πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους όσον αφορά τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας και τις εφαρμοστικές εκθέσεις για το 2013. Συζητήσαμε επίσης και τις εξωτερικές μελέτες. Θα θυμόσαστε ίσως ότι ακόμα τίθεται πρόβλημα όσον αφορά τις εξωτερικές μελέτες με τον προπολισμό του 2012. Παρ' όλα αυτά σχεδιάζουμε ήδη τις σχετικές μελέτες για την επόμενη χρονιά. Οι αποφάσεις θα πρέπει και αυτές να ληφθούν στη συνεδρία της Επιτροπής μας του Δεκεμβρίου. Συνεπώς, οι πολιτικές ομάδες καλούνται στο μεταξύ να σκεφτούν τι εξωτερικές μελέτες μπορεί να χρειαστούμε. Μην ξεχνάτε ότι οι μελέτες αυτές που θα έχουμε μετά το Δεκέμβριο θα έχουν ολοκληρωθεί στα τέλη της επόμενης χρονιάς. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα δηλαδή για τις εξωτερικές μελέτες. Πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε μπροστά. Τι δηλαδή πραγματογνωμοσύνη θα χρειαστούμε στα τέλη της επόμενης χρονιάς. γιατί εξαρτάται από τις νέες πολιτικές που θα έχουμε και τότε εξάλλου θα αξιολογούμε και τις τρέχουσες πολιτικές. Αυτές είναι λοιπόν οι αποφάσεις των συντονιστών. Ωραία, είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία ή να περιμένουμε μέχρι τις 9.30, γιατί 9.30 προβλέπεται η ψηφοφορία. Τι λέτε. Ωραία, σταματάμε, παύση λοιπόν, μέχρι τις 9.30, να αρχίσουμε ακριβώς τις 9.30 της ψηφοφορίες παρακαλώ.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 Constanza, what is, what is the, the... Constanza, η πολιτική σου ομάδα τι άποψη Όψη έχει η πολιτική σου ομάδα για την, για το τελευταίο, για την τελευταία σύνοδο κορυφή. But it's because they, I'm sorry. Because...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 σαν το Αγαπητοί συναδελφοί, ξέρω ότι υπάρχουν ε, προβλήματα για να φτάσει κανείς στο κοινοβούλιο. Και εδώ δεν είμαστε όλοι. Κάποιοι λείπουν, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Τι λέτε, να περιμένουμε ακόμα τρία λεπτάκια ή ε, όχι. Λαμπέρ, για πες. Να ζητήσουμε τους αγρότες να φύγουν. Πρώτα. Ή να αρχίσουμε. Ας αρχίσουμε. Δεν ξέρω οι συνάδελφοι τι λένε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε. Αρχίζουμε με την ψηφοφορία της έκθεσης Μάνκα σε λίγο. Αλλά για να δούμε πώς είμαστε εδώ παρόντες. Μπορούμε να ελέγξουμε πρώτα απ' όλα τις κάρτες σας, να δούμε αν δουλεύουν οι κάρτες σας. Για να ελέγξουμε. Κάντε πως ψηφίζετε κάτι με τις κάρτες σας για να ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. 30 μόνο. 31. Έχουμε απαρτία. Μπορούμε να ψηφίσουμε με 31 ψήφους, έχουμε απαρτία. Ψηφίζουμε λοιπόν. Πέρα της ψηφοφορίας και αρχίζουμε τώρα με το σχέδιο γνωμοδότησης όσον αφορά την βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε για την τροπολογία 9. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρες τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 18-13. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Κατά τμήματα πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, καταπίπτει. Συγγνώμη. 18 τότε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 κατά τμήματα ψηφοφορία υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά αποχές απορρίπτεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία τώρα, ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 30 ψήφους υπέρ. Έκθεση Ρώσα Στεράς Φεραγκούτ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Ας αρχίσουμε την ψηφοφορία. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αυτή. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ κατά. Ας επαληθεύσουμε, τροπολογία 7, αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος, απορρίπτεται με 14 υπέρ 21 κατά. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Για την 14 υπάρχει και μια προφορική, υπάρχει κανείς που ενίσταται, όχι, ωραία. Όπως τροποποιείται λοιπόν, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 17 υπέρ κατά Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει. Τέλος. Και απορρίφθηκε 16 υπέρ 19 κατά. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Ας την επαληθεύσουμε. 20. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος και απορρίφθηκε 16-19. 21 υπέρ. Κατά. Δεν μπορώ να είμαι βεβαία. Ας επαληθεύσουμε την 21. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Και απορρίφθηκε με 14-21. Τροπολογία 22. Εδώ υπάρχει μια ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Α επαληθεύσουμε το δεύτερο τμήμα. Τέλος. Και εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχέ απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχέ απορρίπτεται. 25 υπέρ. Επαλήθευση της 25 αρχίζει. Τέλος. Απορρίφθηκε 14-23. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται λέει η πρόεδρος. Απορρίπτεται. Για την 28 έχουμε... 27 λοιπόν απορρίφθηκε. 28 έχουμε προφορική τροπολογία του κύριου Τεσέρα. Να αντικατασταθεί financial instruments από τις λέξεις funding instruments. Υπάρχει κανείς αντίθετος. 28 λοιπόν όπως τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Τα recital τροπολογία 1 υπέρ κατά επαληθεύουμε. Τροπολογία 1 στις αιτιολογικές σκέψεις. Αρχίζει. Τέλος. Απορρίπτεται με μια ψήφο διαφορά 17-18. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Αρχίζει. Τέλος. 36 υπέρ καμία κατά και μια αποχή. Συγχαρητήρια. Και προχωρούμε στην κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα για τον οδικό χάρτη για την ενέργεια. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Ας επαληθεύσουμε όμως. Τροπολογία 12. Αρχίζει. Και εγκρίνεται. 20 προς 17. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Α, με συγχωρείτε. Εκεί υπάρχει όμως στην συμβαστική 4 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο υπέρ κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής 4. Αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται με 21 υπέρ 16 κατά. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Υπάρχει κανείς που ενίσταται. Κανείς. Ψηφίζουμε όπως τροποποιήθηκε. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Θα σε παληθεύσουμε την 20. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Και εγκρίνεται με 24 ψήφους έναντι 13. 21 υπέρ, κατά. Ας επαληθεύσουμε γιατί το Λαϊκό Κόμμα δεν σηκώνει καλά τα χέρια. Δεν είμαι βεβαία ότι σε ακολουθούν οι συναδελφοί σου Λαμπέρ. Φαντάζομαι να μην, να μην σε ακολουθούμε. Καλά. Εγκρίνεται λοιπόν 24-13 και η τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά πάλι αρχίζει. Τέλος. 31 λέει η πρόεδρος και μία και μία. Now we go for... Θα προχωρήσουμε τώρα στον κύριο Κοζολίνο για το Urban Redevelopment. Τροπολογία 9, υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 10, υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Η 11 έχει αποσυρθεί. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Για την 19 τώρα υπάρχει μια προφορική. Υπάρχει κανείς που ενίσταται. Όχι. Τροποποιείται λοιπόν. Άρα υπέρ 19 εγκρίνεται.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 εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στις citations. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογικές σκέψεις τώρα Τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 20. Υπάρχει εδώ μια προφορική τροπολογία. Αν κανείς δεν ενίσταται τότε ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66. Υπάρχει και εδώ μια προφορική τροπολογία. Αν δεν ενίσταται κανείς ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για την 7. Εδώ επίσης υπάρχει προφορική τροπολογία, αν κανείς δεν ενίσταται, κανείς, καλά, ψηφίζουμε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά παρακαλώ, αρχίζει. Τέλος. 36 υπέρ και μία αποχή. Θαυμάσια. Συγχαρητήρια. Τώρα πάμε στην ε, απονομή συμβολέων ε, παραχωρήσεων, συμβάσεων παραχωρήσεων, Χάιντε Ρουίλε. Υπάρχει μια πρόταση απόρριψης της πρότασης για οδηγία. Να ψηφίσουμε πρώτα αυτό. Ποιος είναι υπέρ αυτής της πρότασης, του να απορρίψουμε την οδηγία. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αυτή η υπόδειξη, αυτή η πρόταση. Άρα θα πρέπει δυστυχώς να ψηφίσουμε. Πρώτη τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρία. Υπέρ. Την ελέγχουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 18 με 18. Ισοψηφία. Απορρίπτεται όμως. 4 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 5 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 6 υπέρ. Ελέγχουμε την 6. Αρχή ψηφοφορίας. Τέλος ψηφοφορίας. Πάλι τα ίδια, 18-18 ισοψηφία. Απορρίπτεται και αυτή. 8. Μιλάμε για τις ε, αιτιολογικές σκέψεις πάντα, έτσι. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 9. Υπέρ, κατά, την ελέγχουμε. Ψηφίζουμε. Δεν μας αναγκάσουμε και να ψηφίσετε. Ε. Τέλος της ψηφοφοριες 17 17-17 απορρίπτεται και αυτή. 10 υπέρ κατά ελέγχουμε τη 10 ψηφίζεται ε, τέλος ψηφοφορίας υιοθετείται αυτή 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά Ελέγχουμε τη 12. Ψηφίστε τώρα. Δεν ψηφίσατε. Τώρα τελειώνει η ψηφοφορία. Υιοθετείτε αυτή. 14. Υπέρ. Την ελέγχουμε. Ψηφίσατε παρακαλώ. Τελειώνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Υπέρ της 15. Κατά. Πάλι δεν ξέρω, πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά το 15. Υιοθετείτε. 16 υπέρ. Υπέρ της 16. Κατά. Την ελέγχουμε και αυτήν. Ψηφίστε. Τέλος ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. 17. Υπέρ. Κατά. Ποχές. Υιοθετείτε. 18. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Ελέγχουμε το πρώτο τμήμα. Ψηφίστε τώρα. Τέλος ψηφοφορίας. υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 19 υπέρ. Συγγνώμη, ξέχασα στην 18, στο δεύτερο τμήμα, υπήρχε και μια προφορική τροπολογία. Ποιος ήταν κατά, υπήρχε κάποιος όχι. Οκ, okay, εντάξει, πέρασε. Κανένας δεν ήταν κατά. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. Πάμε στην 23 υπέρ, την οποία ελέγχουμε. Νομίζω ότι περνάει, αλλά για να δούμε. Υιοθετείτε Με 21-16 υπέρ, 16 κατά. 25 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, 29 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, 30 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 34 υπέρ. Κανένας δεν σηκώνει τα χέρια από εκεί. Τι γίνεται, να ελέγξουμε 34 υπέρ. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 18-19 απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε 35. Έναρξη. Λήξη. Υιοθετείτε. 36 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε 36. Τώρα ψηφίστε. Πέρας. Υιοθετείτε. 37 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 38 υπέρ κατά την ελέγχουμε. Τέλος προφορίας. Υιοθετείτε. 40 και 41 υπέρ, είναι ίδιες ψηφίσμα μαζί κατά εποχές, νομίζω ότι περνάνε, 42 υπέρ, κατά, ελέγχουμε τη 42. Υιοθετείτε. 43 υπέρ. Κατά εποχές υιοθετείτε. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά να ελέγξουμε τη 46 γιατί αν δεν είμαι σίγουρη θα έχω θυάλτες το βράδυ τέλος της χωρίς υιοθετείται 48 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 49 υπέρ να την ελέγξουμε, 49. Τώρα ψηφίστε. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. 18-20. 50 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε αυτή την τροπολογία. Ψηφίστε τώρα. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 17-19. 52 υπέρ. Ίδια κατάσταση. Μπορούμε να ελέγξουμε την 52. Ψηφίστε τώρα. Τέλος ψηφοφορίας. 19-19. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 54 υπέρ. Κατά την ελέγχουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Ελέγχουμε την 56. Ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 57. τελος προφοριας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 18-20. 58 υπέρ. Η ίδια κατάσταση, αλλά σε ελέγξουμε. Τέλος προφορίας Απορρίπτεται. 59. Ίδια κατάσταση. Την ελέγχουμε κι αυτή. Ψηφίστε τώρα. Τέλος. Απορρίπτεται 18-20. 60 και 61. Η 61 έχει αποσυρθεί. Αυτό λέει ο κατάλογος μου. Ναι, μου το επιβεβαιώνετε. Άρα ψηφίζουμε την 60. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Ελέγχουμε την 60. Τέλος ψηφοφορίας. 20-18 περνάει. 62 υπέρ. 62 υπέρ. Κατά. Νομίζω υιοθετείτε. Όχι. Ε. 62 σας αναγκάσα να, να την ελέγξουμε τελικά με αυτά που είπα. Ψηφίστε τώρα. 18-20 απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά έλεγχο 63 ψηφίστε. Τέλος ψηφοφορίας. 19-19 ισοψηφία απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά την ελέγχουμε κι αυτή. Ψηφίστε. Πέρας. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 66 υπέρ. Ελέγχουμε την 66. Τέλος. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείται. 69 υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείται. 70 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 70. Απορρίπτεται. 73 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ελέγχουμε. Την 74. Υιοθετείτε. 75 υπέρ. Κατά. Η κατάσταση ελέγχουμε. 75. Υιοθετείτε. 77 υπέρ. Α, πήδηξα την 76, συγγνώμη. Να ψηφίσουμε την 76 πρώτα. Εσύ τα καταψηφίσεις όλα, Λάμπερ. Τι σε νοιάζει. Ποια λέω. 76, μπας περιπτώσει. Ελέγχουμε την 76. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Πάμε τώρα στην 77. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οι 71 και 72 είχαν αποσυρθεί. Δεν το ήξερε η γραμματεία, γιατί δεν τις ψηφίσαμε. Έχουν όντω αποσυρθεί, έτσι δεν είναι. Κάνουμε τώρα την τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίστε τώρα. Πέρα ψηφοφορίας. 34 υπέρ. Περνάει άνετα. Πάμε στον Derek Vaughan στην έκθεσή του. Δεν είναι εδώ εισηγητής, από ό,τι βλέπω. Ξεκινάμε τη ψηφοφορία. Συμβασμό 1 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμό 2 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμό 3 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμό 4 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμό 11 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 14 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Τροπολογία 10 υπέρ. Την ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 21 κατά, υιοθετείτε. 11 υπέρ, κατά, Νομίζω η ίδια πλειοψηφία, αλλά την ελέγχουμε. Τέλος ψηφοφορίας. 21-21 απορρίπτεται. Συμβιβασμός 5 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 6, συμβασμός 6 δηλαδή υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 7 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 19 υπέρ, Όχι, καταπίπτει. Κοιμάμαι ακόμα. Συμβασμό 8. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Τροπολογία 22. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 9. Συμβασμό 9. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Τροπολογία 27. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 28. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 29. Υπάρχει προφορική τροπολογία. Κάποιος είναι κατά της προφορικής. Όχι. Ψηφίσουμε την 29 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 30 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 10 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 12 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 13 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 39 όπως ε, τροποποιήθηκε προφορικά, κάποιος κατά όχι, ψηφίζουμε λοιπόν ολόκληρο, υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 43 τώρα. Ναι, που όπως τροποποιήθηκε προφορικά, κάποιος κατά της προφορικής τροπολογίας όχι, ψηφίζουμε την αλλαγή υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 15 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 50 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 16 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 53 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Αιτιολογικές σκέψεις. Δεν τις ψηφίζουμε. Πάμε στις υποδείξεις άλλων επιτροπών. Τροπολογία 1 υπέρ κατά. Ελέγχουμε αυτή την πρώτη τροπολογία της Επιτροπής ΕΜΠΛ, Πασχόληση, δηλαδή. Ψηφίστε τώρα. Πέρας, υιοθετείτε. Δύο. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται τρία υπέρ. Την ελέγχουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. 4 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε. 6 υπέρ. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. υιοθετείτε. 7 υπέρ. Ελέγχουμε την 7. Ψηφίζουμε τώρα. Τέλος. Υιοθετείτε. 8. Σε δύο τμήματα. Το δεύτερο καταπίπτει. Ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο μόνο. Υπέρ του πρώτου τμήματος ποιος είναι. Κατά. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της πρώτης τροπολογίας. Της τροπολογίας 8, συγγνώμη. Τέλος ψηφοφορίας υιοθετείται. 9. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι υιοθετείται, αλλά την τσεκάρουμε. Ψηφίστε τώρα. Τέλος ψηφοφορίας. Υιοθετείτε όντως 15 υπέρ κατά αποχές ίδια πλειοψηφία. Υιοθετείτε 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές νομίζω ίδια πλειοψηφία πάλι άρα υιοθετείτε 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ διαφορετική είναι αυτή, να την ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε τώρα. Κλείνει. 22-20 υιοθετείται. 21 υπέρ. Την ελέγχουμε και αυτήν ηλεκτρονικά. Τώρα ψηφίστε. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά τωρα ψηφιζετε απορριπτεται 22 Απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ψηφίστε τώρα. Πέρας ψηφοφορία 42. Τέλεια. Συγχαρητήρια. Και τώρα πάμε σε μια, σε μια πολύ μεγάλη ψηφοφορία. Λαμπέρτ Φανίστερο και Κωνσταντσε Άγγελα Κρέλ. Πρόκειται για τις κοινέ διατάξεις σε σχέση με την ε, εντολή που ψηφίσαμε τον Ιούλιο. Αρχίζει η ψηφοφορία. Περιμένω εδώ να αλλάξει η γραμματεία. γιατί πρέπει να τους έχω εδώ να μου λένε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε αυτή την περίεργη ψηφοφορία γιατί ξεκινάμε με μια ψηφοφορία μπλοκ, ομαδικά δηλαδή. Πρέπει να σας το διαβάσω, είναι... Όχι, δεν χρειάζεται. Τροπολογίες 1 με 26 συμβαστικές, έτσι, τις ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Και πάμε στην τροπολογία 847, στη σελίδα 3, έτσι, 847, πίπερ, βεμπερνίμπλερ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 848, είναι ίδια με την ε, απασχόληση 96 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 851 που είναι ίδια με την 97 της απασχόληση. υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 41 γυναικών υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 852 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόλησης 98 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα πάμε στη σελίδα 6. Τροπολογία 860. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σελίδα 12 τώρα. Τροπολογία 886. 886 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Οχτώ ήτανε. Το ίδιο έχετε όλοι μπροστά σας. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Η γραμματεία τα ίδια έχει στείλει σε όλους αν τα αλλάζουν οι πολιτικέ ομάδε μετά, αυτό δεν είναι δικιά μου θέμα. 886 λοιπόν στη σελίδα 12 ήμασταν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 884 υπέρ, κατά, απόχέ απορρίπτεται. Πρέπει να ψηφίσουμε την 885 τώρα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Σελίδα 17 τώρα. Τροπολογία 97. Υπέρ. Κρέλ και Φανίστερόι. Σελίδα 17. Τροπολογία 97. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 903. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Κοντ 24, που είναι ίδια με την Ήτρα 62. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 907 στην ίδια σελίδα. 907. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 908 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 909 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 912 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 914 είναι ίδια με την κόντι 25 και την ήτρε 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 915 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Κοντ 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήτρε 64 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Επόμενη σελίδα, σελίδα 21. 918 και 921 που είναι ίδιες. Τις ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 920 ίδια με την κόντ 27, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 922, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Κοντ 28, υπέρ, Α, καταπίπτει. Μια στιγμή, μια στιγμή. Πρέπει να είμαστε σίγουροι. Καταπίπτει, ναι. Η Ήτρε 65. Όχι, λοιπόν, ψηφίζουμε. Ήτρε 65 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πάμε τώρα στη σελίδα 24. Ψηφίζουμε την τροπολογία 929. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Σελίδα 26 τώρα. Τροπολογία 1142. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1143 τώρα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συνεχίζουμε και πάμε στη σελίδα 34. Εδώ έχουμε μία συμβιβαστική τροπολογία που δεν αποτελούσε μέρος του, της ομάδας που ψήφισαν πριν, 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 27. Επόμενη σελίδα, κοντ 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, 4 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόλησης 1. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Γυναικών 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προπολογισμών 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προπολογισμών 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προπολογισμών 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προπολογισμών 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προπολογισμών 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εικόν 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οίκον 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 28. Στην αντιλογική σκέψη 5. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ένα στην επόμενη σελίδα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ κατά αποχές NV2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σελίδα 41 τώρα 193 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 30 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στο δεύτερο τμήμα της 194. 194 δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 197 δεύτερο τμήμα πάλι. 197 δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 στην επόμενη σελίδα. 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 202. 202 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 204 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τραν 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμών 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 31 τώρα στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 48 τώρα. Ήτρε 1. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 213. Υπάρχει προφορική τροπολογία. Είναι κανείς κατά. Ωραία, ψηφίζουμε τότε την τροποποιημένη τροπολογία. Υπέρ, κατά. Ξανά μια στιγμή, γιατί... Ε, ναι, υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται με την προφορική τροποποίηση αυτή. Τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 32 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα, γυναικών 4. Φαμ 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήτρε, α, όχι μάλλον, συμβαστική τροπολογία 33 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σελίδα 55 τώρα, συμβαστική τροπολογία 34, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σελίδα 59. Είναι επόμενη συμβαστική τροπολογία 35. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άγκρι 5, εικόν 3, γυναικών 5, 235, 236 είναι ίδιες και οι 237. Τις ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 10. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Εξήντα τρία και εικον τέσσερα υπέρ Σελίδα 63, έτσι, εικόν 4 κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε, έξι όχι. Συμβαστική τροπολογία 36 τώρα. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 37 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα, 248 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 250 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 251 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 252 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οίκον 5, καταπίπτει. Ήτρε 7, την ψηφίζουμε. Ήτρε 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 38 και υπάρχει και προφορική τροποποίηση της Κωνσταντσα Κρέλ και του Λαμπέρ Φανίστερο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ποιος θα μας την παρουσιάσει. Ή την ξέρουν. Α, την ξέρει ο κόσμος, εντάξει. Είναι κανείς κατά της ε, προφορικής τροποποίησης. Α, υπάρχει κάποιος που είναι κατά. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ψηφίσουμε την ε, προφορική τροποποίηση, αλλά την αρχική τροπολογία. Συμβαστική τροπολογία 38, λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 254 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 256 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πρέπει κάτι να ελέγξουμε μια στιγμή. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία κοντ 6. Σελίδα 66. Ε. Κοντ 6. Και ήτρε 8 είναι ίδιες. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. αποχέ, απορρίπτονται. Εκόν 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 260. Υπέρ. Κα... Υπέρ. Κατά. αποχέ, απορρίπτεται. Συμβαστική 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 261 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 262 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε στην επόμενη σελίδα 265. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άγκρι 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 42 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 267 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. απασχόληση 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ένβιδε 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 271 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κοντ 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήτρε 10 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σελίδα 73, τροπολογία 280. Α, όχι. Η 47 μου ξέφυγε. Συμβαστική τροπολογία 47 πρώτα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στη 280. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 285 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 76 σελίδα πάμε τώρα. Τροπολογία 296. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι επόμενες καταπίπτουν. 293. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εκόν 9. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 297 κατά πίπτη, 53 τώρα, συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απασχόλησης 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Γυναικών 8 όχι, δεν την ψηφίζουμε αυτή. Τις ε, προπολογισμών 18, απασχόληση 14, ήτρε 12 κλπ. κλπ. Όλες αυτές είναι ίδιες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 54. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 80, 314 τροπολογία υπέρ να περιμένουμε λίγο. Ωραία, σελίδα 80, τροπολογία 314. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Κοντ 11, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. «317 τώρα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 55 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 300... Όχι. Συμβιβαστική 56 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα τώρα, τροπολογία 57 συμβαστική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 320 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. NV7 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Επόμενη σελίδα. Συμβαστική 58. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, πες 3 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Πασχόλης 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 326 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 329 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένβη 8 σελίδα 86. Ένβη 8 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 64 υπέρ, κατά απόχέ εγκρίνεται. 65 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκόν 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και πάμε τώρα στη σελίδα 90. Σελίδα 90. Κοντ 14 και Ήτρε 15. Σελίδα 90. Κοντ 14 και Ήτρε 15. Τι ψηφίζουμε υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 68 τώρα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Σελίδα 92 έχουμε τη συμβαστική 69. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 94 συμβαστική 70. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και συμβαστική 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πρέπει να σας ρωτήσω. Δεχόμαστε τις τροπολογίε αυτές που ψηφίσαμε για να συνεχιστεί η διαπραγματεύση στο Συμβούλιο. Θυμόσαστε ότι και τον Ιούλιο σας ε, το είχα ρωτήσει. Έτσι, αυτή είναι η εντολή. Δεχόμαστε λοιπόν ως εντολή αυτά τα οποία μόλις ψηφίσαμε για να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Δεν βλέπω να αντιτίθεται κανείς. Πρέπει να, το να ψηφίσουμε τώρα. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Ομόφωνα το δεχόμαστε δηλαδή ως εντολή. Δεχόμαστε αυτή την εντολή, έτσι. Καλώς. Έχουμε άλλη μία ψηφοφορία όμως αγαπητοί συνάδελφοι του Μάρκος Πίπερ. Έτσι. Θα θυμόσαστε ίσω ότι τον Ιούλιο δεν τα ψηφίσαμε όλα γιατί ορισμένα εξαρτώνταν από την εντολή. Τώρα λοιπόν έχουμε την υπόλοιπη εντολή και άρα μπορούμε να ψηφίσουμε τα υπόλοιπα τμήματα της έκθεσης του Μάρκου Σπίπερ και ξεκινάμε με τη συμβαστική 5. Υπέρ. Λαμπέρ. Το λέω για σένα, συμβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. Τροπολογία 78 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. 79 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. Συμβασμό 9. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 111. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 116. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 123. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 124. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 126 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14 υπάρχει προφορική τροπολογία του εισηγητή, κατά, της προφορικής κάποιος, όχι. Ψηφίζουμε την 14 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 132, όχι, καταπίπτει. Πάμε στο 18, υπέρ. Να την ελέγξουμε εκτονικά Τέλος. 24.16 Συμβασμός 2. Για τις αιτιολογικές σκέψεις. Υπέρ, κατά, αποχές. Υιοθετείτε. 37 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά, κατά αποχές υιοθετείται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε τώρα. τη ψηφοφορία. Υιοθετήσαμε την έκθεση του Μάρκου Πίπε Συγχαρητήρια. Μάλιστα έχουμε τελειώσει νωρίτερα από ό,τι προβλέπαμε. Αλλά να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας της διάταξης που είναι μια έκθεση της για την επίσκεψη της αντιπροσωπείας Ρέγγι. Ποιος είναι έτοιμος να παρουσιάσει την έκθεση. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, λέει ο κύριος Ματούλα. Μπορώ να σας παρουσιάσω την έκθεση. για την ε, αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ρέγγι που πήγε στη συνοριακή περιοχή ε, μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, Languedoc-Roussillon και Καταλωνία. Στις 29 με 31 Οκτωβρίου του 12 έγινε αυτή η επίσκεψη. Από την αρχή θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι εγώ προσωπικά νομίζω ότι ο προορισμός ήταν πολύ ωραία επιλεγμένος δεδομένης της παράδοσης που υπάρχει για τη συνοριακή συνεργασία στις περιοχές αυτές. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες συνεργασίας στα γαλλο-ισπανικά σύνορα. Με βάση την αρχή της εδαφικής συνεργασίας και της, ε, πολιτικής, ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής. Υπάρχουν πολλές διμερείς συμφωνίες και πολλές ε, ισχύουν εδώ και πολλά χρόνια. Η συνοριακή περιοχή που επισκεφτήκαμε στα πλαίσια της εδαφικής συνεργασίας και του στόχου για την εδαφική συνεργασία προωθεί προγράμματα με σκοπό την συνεργασία για την καινοτομία, το σχεδιασμό της συνεργασίας, την ενίσχυση των διασυνοριακών δικτύων, την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η επίσκεψη ξεκίνησε στις 29 Οκτωβρίου, όπως σας είπα, μια Δευτέρα στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Βαρκελόνη, όπου μας ενημέρωσαν για το τι κάνουν οι Ισπανοί στα πλαίσια του προγράμματος και της συνεργασίας και συνεχή συνεχεία αντιπροσωπεία επισκέφτηκε ένα νοσοκομείο στην Ισπανία που είναι ένα πρωτοποριακό διασυνοριακό νοσοκομείο, ένα από τα πρώτα της Ευρώπης. Είναι σε μια ορεινή περιοχή και, προβλέπει, και παρέχει υγειονομική υπερίθαλψη σε 30.000 άτομα, τα οποία ζουν εν γέννη σε απόμακρες ορεινές περιοχές και το χειμώνα η περιοχή έχει επιπλέον 150.000 κατοίκους ως αποτέλεσμα των, ε, του τουρισμού για χειμερινά αθλήματα κτλ. Τουρισμός δηλαδή ουσιαστικά. Υπάρχει το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που χρηματοδοτεί κυρίως αυτά τα προγράμματα το πρόγραμμα αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί δίνει υγειονομική περίθαλψη όχι μόνο στον τοπικό πληθυσμό αλλά και στους τουρίστες αυτούς που επισκέπτονται την περιοχή το χειμώνα για χειμερινά σπορ, για σκι δηλαδή και άλλα χειμερινά αθλήματα. Πολλές, πολλοί φορείς διασυνοριακοί δημιουργήθηκαν ακριβώς για να παρέχουν ε, ιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες. Αντιμετωπίσαμε κάποιες δυσκολίες ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Υπάρχουν θέματα, υπάρχουν προβλήματα που παρεμποδίζουν τα προγράμματα αυτά. Με ποια έννοια. Δεν υπάρχει δηλαδή ενιαία ε, νομοθεσία για την υγειονομική περίθαλψη στη Γαλλία και στην Ισπανία. Δεν είναι ίδια η νομοθεσία και αυτό μερικέ φορές αποτελεί πρόσκομα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψη στην ισπανική πλευρά των συνόρων είχαμε συναντήσεις με συμβούλους δημοτικούς, περιφερειακούς και με υπουργούς της Ανδόρας, με τους οποίους συζητήσαμε τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών αυτών, δηλαδή Ισπανίας, Γαλλίας, αλλά και της Ανδόρας. Εν συνεχεία επισκεφθήκαμε τη Γαλλία. Στο Περπινιό πήγαμε, πιο συγκεκριμένα, όπου η αντιπροσωπεία παρέστησε ένα πολιτιστικό έτσι, συμβάν, ένα θέατρο που χρηματοδοτείται από το Interreg και που προωθεί τον τις διαπολιτιστικές εκδηλώσεις και μια μεγαλύτερη κοινωνική ανοχή. Συζητήσαμε με τις τοπικές αρχές και με τον δήμαρχο του Περπινιό μάλιστα, ο οποίος συμμετείχε, και με τον Περιφερειάρχη. Συζητήσαμε επίσης τη διασυνοριακή συνεργασία μαζί τους στον τομέα των τεχνών, του θεάτρου, Ο πολιτιστικός τομέας θα παραμείνει επιλέξιμος τομέας υπό τα διαρθρωτικά ταμεία, για τα, από τα κονδύλια δηλαδή των διαρθρωτικών ταμείων και, και στο Περπινιό και στη Χερόνα υπάρχει μεγάλη συνεργασία. Όπως είπα, συναντήσαμε εκπροσώπους των τοπικών αρχών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και με μέλη του Πανεπιστημίου του Περπινιό, όπου είδαμε πόσα πολλά προγράμματα υπάρχουν στην περιοχή και τα συζητήσαμε. Εφτά μέλη της Επιτροπής συμμετείχαν σε αυτό το ταξίδι, σε αυτήν την αντιπροσωπεία στη διασυνοριακή περιοχή Γαλλίας-Ισπανίας. Συνολικά είχαμε 25 άτομα στην αντιπροσωπεία, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Γραμματείας και διερμηνής. Η αντιπροσωπεία ανακάλυψε ότι η περιοχή έχει προγράμματα πολύ υψηλής ποιότητας και οι τοπικές αρχές χάρηκαν που πήγαμε εμείς εκεί, ευχαριστήθηκα με την παρουσία μας και από τις συναντήσεις που είχαμε προκύπτει ότι υπάρχει μια προστιθέμενη αξία από αυτές τις συζητήσεις και για μας αλλά και για τις τοπικές αρχές. Οι άνθρωποι που συναντήσαμε μίλησαν για την ανάγκη για περισσότερα κονδύλια για τη διασυνοριακή συνεργασία και ανακαλύψαμε και φαντάζομαι και άλλοι συνάδελφοι θα το σχολιάσουν αυτό το θέμα, ότι υπάρχει ένα μέσο που έχει τεράστιο δυναμικό. Η Ευρωπαϊκή Όμιλη Εδαφικής Συνεργασίας, όπως λέγονται. Πολλοί με τους οποίους μιλήσαμε είπαν ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Όμιλη είναι ένα πολύ επιτυχημένο μοντέλο. Είπαν ότι είναι ένα από τα λίγα ευρωπαϊκά νομοθετικά πλαίσια που πραγματικά έχει τεράστια επιτυχία. Υπάρχουν 280 τέτοιοι όμιλοι στην Ευρώπη και από αυτούς οι πέντε είναι στα γαλλοϊσπανικά σύνορα. Οι ευρωβουλευτές που συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία είδαν πώς αναπτύσσονται, πώς εξελίσσονται τα προγράμματα σε αυτή τη συνοριακή περιοχή και είδαμε το τεράστιο δυναμικό που υπάρχει στην εδαφική συνεργασία και στους ευρωπαϊκούς όμιλους εδαφικής συνεργασίας. Είδαμε πραγματικά τι γίνεται εκεί στην περιοχή ε, και αποφασίσαμε ότι πραγματικά έχει νόημα η συνέχιση της χρηματοδότησης στον τομέα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη που συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία και όχι μόνο αυτούς, αλλά και τη γραμματεία, τους τεχνικούς και τους διερμηνείς. Η επίσκεψη ήταν πολύ καλά οργανωμένη, ήταν μια μεγάλη επιτυχία, δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα και νομίζω ότι ήταν πολύτιμη εμπειρία και για μας, αλλά και για τις τοπικές αρχές με τις οποίες συναντηθήκαμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαρή Τερέζ Σάντσε Σμιτ, που ήταν ε, αυτή που μας είπε αυτή την ιδέα να επισκεφτούμε αυτή την όμορφη περιοχή. Η Μαρή Τερέζ ε, ήταν πάρα πολύ έτσι, ζεστή η κοδέσπινα και μας βοήθησε πάρα πολύ σε όλα τα μέρη που επισκεφτήκαμε. Έτσι μας έδωσε ωραίες συμβουλές. Καλό τους συναδέλφους να δουν τα έγγραφα τα οποία συντάξαμε μετά την επίσκεψη και να μιλήσουν στους ευρωβουλευτές που συμμετείχαν στην επίσκεψη αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συναντήσαμε που ήταν πάρα πολύ ζεστοί απέναντί μας και μας δέχτηκαν μεγάλη θέρμη. Ε, δεν ήταν πάντα όμως όλα ωραία και καλά, γιατί μια φορά σε μια επίσκεψη από τους 22 βαθμούς πέσαμε στους μείον 2. Και ο Φράντσες Κοντάντζελη, ο κ. Ντεβόν, η Ρόζα Εστεράς Φεραγκούτη και η Μαρία Γκογιαν Περές. Ήταν μια ολόκληρη ομάδα, δηλαδή δεν ήταν μόνο η Μαρή Τερές. Οι υπόλοιποι θέλουν να προσθέσουν τίποτα. Ο κύριος Τσέλερ, ευχαριστώ και εσάς κυρία Πρόεδρε και τον συνάδελφό μου για την πλήρη παρουσίαση των λεπτομεριών της ε, επισκέψεως. Ευχαριστώ επίσης, έστω και αν είναι απούσα, την Μαριτερές για την προετοιμασία του ταξιδιού, καθώς και την βοήθεια στην εκτέλεση. Σε δυόμιση μέρες μπορέσαμε πραγματικά να ρίξουμε μια βαθιά, ματιά σε βάθος στη ζωή τη περιφέρεια αυτής και αυτό οφείλεται στι προσπαθίε τη. Δυστυχώ το ενδιαφέρον των συναδέλφων όπως και εδώ άρρωστε για την ακρόαση ήταν περιορισμένο διότι ήμασταν μοναχά τέσσερις ε, βουλευτέ από δύο πολιτικές ομάδες. Όταν γίνεται όλη αυτή η προετοιμασία για μια τέτοια αποστολή με μεγάλη προσπάθεια και δαπάνες, τουλάχιστον θα πρέπει η αντιπροσωπεία να αποτελείται από τον μέγιστο αριθμό των ε, βουλευτών. Για μένα η επίσκεψη ήταν σημαντική, διότι όπως είπε και ο Ζωζεφ προηγουμένως, στην μεθοριακή αυτή στη μεθοριακή αυτή περιοχή Ισπανίας-Γαλλίας ήδη υπάρχουν πέντε έργα της διαμεθοριακής αυτής συνεργασίας και μάλιστα και οι παλαιότερες που εξακολουθούν να ε, λειτουργούν. Και όπως ακούσαμε σχεδιάζεται και η ίδρυση και νέων. Γιατί τα ταξίδια βέβαια συμβάλλουν στο να ανοίξει το μυαλό των ανθρώπων. Και εγώ διαπίστωσα ότι σε αυτή, την, σε αυτή τη μεθοριακή περιοχή Ισπανίας-Γαλλίας και πέρα των συνόρων διατηρείται αυτή η καταλανική ταυτότητα των ανθρώπων ε, είδα περισσότερες καταλανικές σημαίες από ε, γαλλικές. Εκεί ισχύει και η διγλωσία, για παράδειγμα στις πινακίδες με τα ονόματα των δρόμων. Και αυτό εδώ και 100 χρόνια. Πολλοί από τους ντόπιου μου είπαν ότι η Βαρκελόνη για αυτούς είναι πολύ κοντύτερα από ότι το Παρίσι. Και γι' αυτό βέβαια θέλουν και να μπορούν να συνεργάζονται στενά και πέρα από τα σύνορα. Τα διαφορετικά, τα διαφορετικά νομικά συστήματα και εκεί, αλλά όπως βλέπουμε ας πούμε και στα γερμανοπολωνικά σύνορα, δεν βοηθούν. Γι' αυτό και αναμένουν τον νέο κανονισμό για τις διαμεθοριακές συνεργασίες, η οποία νομοθεσία θα διευρύνει το νομικό πλαίσιο και θα προσφέρει και μια ασφάλεια δικαίου για την συνεργασία σε διαμεθοριακά έργα. Ο Ζωζέφ ήδη ανέφερε το Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο του Περπινιάου, που επιθυμεί να είναι το πρώτο που θα έχει αυτό το διαμεθοριακό χαρακτήρα. Μέχρι τώρα μπλοκάρει το Παρίσι. Το Πανεπιστήμιο μας είπε ότι εάν μπορούν να βασιστούν σε αυτή τη νέα νομική βάση που θα προσφέρει ο κανονισμός, θα εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα αυτή έτσι ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν δραστηριότητε και στην Ισπανική περιφέρεια που είναι πέραν των συνόρων. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντική όθηση για την εργασία μας το γεγονός ότι μπορέσαμε και επισκεφθήκαμε και είδαμε πώς λειτουργούν τα εργαλεία εντός αυτά τα οποία εδώ εμείς συζητούμε και εγκρίνουμε, πώς διεξάγεται η συνεργασία αυτή πέραν των ορίων των περιφερειών και πέραν των κρατικών σύνορων που εξακολουθούν να υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις ή σχόλια υπάρχουν? Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Μαρία Τερέσα που μας έδωσε την δυνατότητα να γνωρίσουμε από κοντά την διασυνοριακή συνεργασία. Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε δύο πυλώνες που θεωρώ ότι είναι πολύ βασικοί και αυτή είναι η υγεία και η εκπαίδευση το Διασνοριακό Πανεπιστήμιο δηλαδή. Αλλά και το νοσοκομείο είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για το τι πρέπει να είναι η Ευρώπη. Είναι ένα ε, νοσοκομείο πολύ κοντά στα γαλλικά σύνορα, ένα χιλιόμετρο, και όσοι ζουν εκεί γύρω, πολύ πιο εύκολα προσφεύγουν σε αυτό το νοσοκομείο παρά στο Περπινιάν που είναι 80 χιλιόμετρα πιο πέρα και που είναι ένας δύσκολος δρόμος. Συνεπώς, είναι πολύ ενδιαφέρον που υπάρχει αυτό το νοσοκομείο που δεν είναι τόσο για ασθένειες που απαιτούν βέβαια διαφορετικό εξοπλισμό, αλλά πιο πολύ ανταποκρίνονται στις ε, πρώτες ανάγκες του κόσμου. Έχουν ε, εκεί πέρα γυναικολογικό τμήμα, ε, γεννιούνται παιδιά εκεί, φροντίζουν τους ηλικιωμένους κλπ. Με φτύριο δηλαδή. Όλοι Επίσης όσοι έχουν κάποιο πρόβλημα με τα χειμερινά αθλήματα ε, μπορούν επίσης να πάνε στο νοσοκομείο αυτό. Τα 8 εκατομμύρια ευρώ ήταν ευρωπαϊκά κονδύλια. Τώρα η συντήρηση πυρικοδότηση είναι, ανήκουν και στην Καταλωνία και στην ε, Γαλλία. Κάπως κατανέμεται ανάλογα με τον πληθυσμό. Από την άλλη, η εικόνα που παίρνουν ε, οι τουρίστες που πηγαίνουν σε αυτή την περιοχή είναι η εικόνα της Ευρώπης, δηλαδή η εικόνα ενός νοσοκομείου που εξυπηρετεί τους Ευρωπαίους. Και στο Πανεπιστήμιο τώρα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει, του Περπινιά δηλαδή, υπάρχει μεγάλη ε, συνεργασία και έρχονται και φοιτητές και από άλλες χώρες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός. Και υπάρχει και το θέατρο είναι σημαντικός ο πολιτισμός, δηλαδή να μπορούν όλοι όσοι ζουν στην περιοχή να ε, έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τη Μαρία Τερέσα, η οποία ε, μας έδειξε κάτι που βοηθάει. Δεν είναι μόνο το Πουτσερδάτ και το Περπινιάν, αλλά είναι κάτι που αφορά όλους τους Ευρωπαίους, να ξέρετε. Ευχαριστώ και πάλι. Ε, Ευχαριστώ. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι θα πάει αυτή η έκθεση στη διάσκεψη των Προέδρων. Η έκθεση επίσης επιβεβαιώνει την ιδέα ότι το να κάνουμε μια τέτοια στοχοθετημένη επίσκεψη για να διαπιστώσουμε πώς λειτουργεί ένα τέτοιο ευρωπαϊκό εργαλείο είναι χρήσιμο όχι μόνο για την περιφέρεια, αλλά για να δούμε και πώς θα πάει το ίδιο το εργαλείο, αν δηλαδή υλοποιεί τους στόχους της πολιτικής. Τόμα πάμε στο δικό σημείο της ημερήσιας διάταξης, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για την, το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Ο Τόμας Ντόιτς ετοίμασε μία έκθεση ε, για την Επιτροπή Οίκων. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, κυρία Πρόεδρε, να μιλήσω για αυτό το θέμα. Πρόκειται για ένα σχέδιο γνωμοδότησης. Θα ήθελα να κάνω καταρχήν δύο παρατηρήσεις και εν συνεχεία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τρεις σκέψεις, ούτω ώστε να συμπληρώσω το γραπτό κείμενο που έχετε μπροστά σας. Πρώτον, για την ετήσια εξέταση της ανάπτυξης για το 2013, θα θυμάστε την γυναίκα του Κολόμπο, θυμάστε αυτή την αστυνομική σειρά. Ε, συχνά μιλάμε ε, για αυτή την έκθεση, μιλάνε μάλλον στην στη σειρά για αυτή τη γυναίκα, αλλά κανένας δεν την είδε ποτέ. Έτσι είναι και αυτή η, αυτό το κείμενο. Αυτή τη βδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει αυτό το κείμενο. Ακούμε να μιλάνε για αυτό κτλ. αλλά θα το μάθουμε, θα το γνωρίσουμε αυτό το κείμενο τώρα μόλις, ως ο νουπο δηλαδή. Αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε για την Επιτροπή μας όμως. Γιατί θα έχουμε χρόνο για να ετοιμάσουμε τις νομοδοτήσεις μας και τις τροπολογίες μας. Αυτό ήταν το πρώτο που ήθελα να σας πω. Δεύτερον, όταν μιλάμε για την πολιτική συνοχής, καλό και άγιο αυτό αλλά μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για αυτή την πολιτική, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τι έγινε στο τέλος της ε, περασμένης εβδομάδα στην Σύνοδο Κορυφής. Δηλαδή τι συνέβη και τι δεν συνέβη, για να το πω καλύτερα, σε σχέση με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτή είναι η δεύτερη σκέψη. Η τρίτη σκέψη. Φυσικά η ετήσια εξέταση της ανάπτυξης στο σχέδιο του κειμένου μου εστιάζεται στην πολιτική συνοχής και στο ρόλο αυτής της πολιτικής στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι πεπισμένος ότι αν έχουμε φιλόδοξες πολιτικές επενδύσεων και αλληλεγγύης και αν η πολιτική συνοχή χαρακτηρίζεται από το επίθετο φιλόδοξος, τότε θα έχουμε όλα τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε την κρίση τα επόμενα χρόνια. Και όπως λέω και στο κείμενό μου, στο σχέδιο γνωμοδότησής μου, θα πρέπει, ότι, θα πρέπει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πολιτικής συνοχής να μην υποστεί δραστικές περικοπές. Νομίζω ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να είναι ευέλικτη πολιτική, ούτως ώστε να βοηθάει τις περιφέρειες στη διαχείριση της κρίσης. Θα να σας πω λοιπόν ότι αναφέρω με κατ' επανάληψη ε, στο πρόβλημα της μείωσης της ε, συγχρηματοδότησης στο κείμενό μου. Σε ό,τι αφορά τώρα την απορρόφηση των κονδυλίων του, των Ταμείων Συνοχής, θα πρέπει να έχουμε εθνικούς προπολογισμούς υγιείς, στέρεους και που θα περάσουν από διορθωτικές μεταρρυθμίσεις. Η σταθερότητα των εθνικών προπολογισμών είναι σημαντικό και είναι σημαντικές οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επίσης ε, γίνεται αναφορά με έμφαση σε αυτό το σημείο. Η κρίση είναι πολύ σημαντική, προκαλεί ανεργία στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν η προσέγγιση μου ήταν να τονίσω την ε, στρατηγική Ευρώπη 2020. Έχουμε το στόχο το 75% των ατόμων 20 με 64 χρονών να έχουν μια δουλειά. Είναι πολύ εφιλόδοξο αυτό. Αυτό σημαίνει δημιουργία θέσεων απασχόληση. Σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν οικονομικέ πολιτικέ υπέρ τη ανάπτυξη για να στηρίξουμε τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, να την προωθήσουμε αυτή. Μάλιστα. Συνολικά μπορώ να σας πω ότι χρειαζόμαστε μια πολιτική συνοχής σταθερή που να έχει την απαραίτητη χρηματοδότηση. Αυτό το τονίζω στο σχέδιο γνωμοδότησής μου. Εν ώψη της ετήσιας εξέτασης για την ανάπτυξη για το 2013. Αυτά ήθελα να σας πω. Θέλετε να ρωτήσετε τίποτα. Ε, α, ναι, εγώ, η κυρία Κλέβα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ντόιτς για την έκθεση που συνέταξε με ιδιαίτερα καλό τρόπο. Έχω και εγώ το πρόβλημα ότι συνέταξα το σχέδιο γνωμοδοτήσεως για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τα κοινωνικά θέματα δηλαδή από το 2013 και μετά. Δεν έχω το κείμενο. Αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται. Υποθέτουμε. Υποτίθεται ότι την εβδομάδα θα λάβουμε το κείμενο. Και Νομίζω ότι και για αυτό το θέμα και για το επόμενο της ημερήσιας διαταξής μας, τα κείμενα που συντάσσουμε θα μπορέσουν να βελτιωθούν και να τροποποιηθούν. Γενικά, συμφωνώ με τον εισηγητή, ο οποίος απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Είναι ακριβώς οι δύο στόχοι που προσπαθούμε να επιτύχουμε το δυνατόν συντομότερο. και αυτά αποτελούν την πραγματική πλατφόρμα που σε αυτήν πρέπει να στηριχτούμε για να κάνουμε την κατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού. Η δική μας Επιτροπή πρέπει να εκφράσει την άποψη ότι η πολιτική συνοχή είναι ο βασικός μηχανισμός για ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά συζητούνται και, στο, και στη διάσκεψη κορυφής Εκτός αυτού, θα υποβάλω βέβαια και άλλα σχόλια αργότερα και τις τροπολογίες μου για την έκθεση του κυρίου Ταμάς Ντόιτς. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ταχθεί υπέρ μιας μεγαλύτερης και βαθύτερης νομιμότητας των διαδικασιών μας, ξεκινώντας από την ετήσια επιθεώρηση ανάπτυξης, για την οποία έχουμε μιλήσει και την οποία έχουμε ζητήσει πολλές φορές, επ' αυτού πρέπει να επιμείνουμε, η διαθεσμική διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να γίνει διαφανέστερη και πρέπει να οδηγήσει σε περισσότερες ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές που θα βασιστούν στις παλαιότερες για να στηρίξουν τις νέες αιτήσει επιθεωρήσεις για την ανάπτυξη. Δεν υπάρχει όμως διασύνδεση μεταξύ των guidelines του περσινού χρόνου και των φετινών. Πρέπει να φωτίσουμε και τις αρνητικές επιπτώσεις, καθώς και να τονίσουμε το αποτέλεσμα spillover, δηλαδή ότι κάποια πράγματα πηγαίνουν και αλλού, ξεφεύγουν και πηγαίνουν και αλλού. Και να διορθώσουν τα προβλήματα οι χώρες μέλη προβλήματα δηλαδή για τα οποία δεν φέρουν την ευθύνη. Το τρίτο θέμα που με απασχολεί είναι το ελάχιστο επίπεδο κοινωνικής προστασίας και των σχετικών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή. Οι συλλογικές συμβάσεις και διαπραγματεύσεις και συμβάσεις δηλαδή στις χώρες μέλη αποτελούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Το τελευταίο θέμα που συζητούμε στην Επιτροπή μας είναι ότι η πολιτική συνοχή είναι πολιτική επενδύσεων, επενδύσεων στην απασχόληση, σε καινούριε δουλειές. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ποινές στις ε, περιφέρειες λόγω της μακροοικονομικής τους κατάστασης που οφείλεται ωστόσο στις αποφάσεις των κεντρικών κυβερνήσεων των χώρων μελών. Γι' αυτό και είμαι αντίθετη με οποιαδήποτε επιβολή όρων μακροοικονομικών και αυτά πρέπει να περιληφθούν βέβαια και στην ετήσια επιθεώρηση ανάπτυξης. Μάλιστα, δεν έχω άλλα. Τόμας, θέλετε εσείς να σχολιάσετε. Όχι. Καλά. Αυτό που κρίνεται σήμερα είναι, πρέπει να εγκριθεί μάλλον σήμερα, είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Εγώ προτείνω την Τετάρτη 12 στις 12 το μεσημέρι. Εδώ τέλος πάντων λέει η πριν, πρόμεσημβρινή, εννοείται φυσικά 12η μεσημερι. Και ελπίζω τώρα, αν συμφωνήσουμε, ότι θα γίνει κατανοητό ότι οι τροπολογίες μπορούν να γίνουν μόνο στα αγγλικά. Δεν προλαβαίνω να μεταφραστούν. Αλλά αυτό έχει συζητηθεί ήδη με τις πολιτικές ομάδες καθώς και με τον εισηγητή. Και ως συνήθως όλοι έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε τροπολογίες απευθείας στην Επιτροπή Οικονομικών χωρίς να περάσετε από τη δική μας διαδικασία μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Εδώ λίγη συζήτηση του θέματος αυτού. Ελπίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη ε, γνωμοδότηση της ε, Μόιτσα Κλέβα που νομίζω ότι ήδη στην ουσία την παρουσίασε. Βέβαια, επισήμως πρέπει να περάσουμε και στη δική σας γνωμοδότηση και σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Τα βασικά σημεία της έκθεσής μου. Όπως είπα, το πρόβλημα είναι ότι το έγγραφο θα είναι διαθέσιμο μόλις στα τέλη της εβδομάδος. Με τους σχεώδεις ηγητές είμαι βεβαίως ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο με την κατάθεση τροπολογιών και νέων διατυπώσεων. Διότι εδώ είμαστε... Κάνουμε γνωμοδότηση μάλλον για την Κοινωνική Επιτροπή και Επιτροπή και Απασχόλησης. Και όπως είπα και πριν, μιλούμε για την πολιτική συνοχής ως βασικής πολιτικής επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην απασχόληση στους περισσότερο από άλλες πολιτικές. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να παίξει τον ρόλο της η δική μας Επιτροπή να συντάξει γνωμοδότηση, βέβαια, αλλά λόγω των περιορισμών των χρονικών περιορισμών δηλαδή, καλούμαστε να συντάξουμε ένα κείμενο εκ των προτέρων. Αύριο θα ακούσουμε την ακρόαση του κ. Άντρους. Ελπίζω δε ότι το κείμενο που θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση, για την επανεξέταση μάλλον του 2013, θα είναι πλέον φιλόδοξο του φετινού και ότι θα περιλάβει επανεξέταση και των guidelines για τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει παρόλο που το είχαμε ζητήσει ήδη από πέρυσι. Η πολιτική συνοχής ως η βασική επενδυτική πολιτική θα πρέπει να έχει ως στόχο να μειώσει τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών και να οδηγήσει σε μια αποδοτική και διαρκή ανάπτυξη που θα οδηγήσει και αυτή με τη σειρά της στην απασχόληση. Αυτά τα λέμε βεβαίω εδώ και ένα χρόνο. Δεν είναι τίποτε το νέο. Τώρα τι άλλο έχουμε να πούμε. Είναι σαφέ ότι η πολιτική συνοχή πρέπει να προσαρμοστεί στις περιφερειακές ανάγκες ανά περίπτωση και να μειώσει τι διαφθορτικές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών. Αυτό για μένα είναι σημαντικό. Χαίρομαι για την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την αναδιάθεση μη απορροφηθέντων κονδυλίων υπέρ των μικρών και μεσών επιχειρήσεων και θα πρέπει αυτά να οδηγηθούν σε επενδύσεις για μεγαλύτερη αποδοτικότητα της ενέργειας καθώς επίσης και για την απασχόληση νέων. Και ελπίζω η Κομισιόν να ζητήσει από τις χώρες να χρησιμοποιήσουν πλήρως τα κονδύλια των διαθροτικών ταμείων για να καταπολεμήσουν την μακρόχρονη και διαρθρωτική ανεργία. Η Κομισιόν ανακοίνωσε ήδη ότι θα υποβάλει πρωτοβουλία για την εγγύηση υπέρ της νεολαίας, Youth Guarantee, και αυτό αναφέρεται και στη γνωμοδότηση. Αλλά η ανακατανομή μη απορροφηθέντων κονδυλίων νομίζω ότι αποτελεί και το κλειδί εδώ για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Άλλος κανείς, λέει η Πρόεδρος, εκ των σκιωδών εισηγητών ή εσείς τα μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου δύο μικρές παρατηρήσεις. Έχουμε δύο γνωμοδοτήσεις που μοιάζουν η κυρία Κλεβά έχει κάνει μια πολύτιμη δουλειά. Τρία πραγματάκια θα ήθελα να συμπληρώσω. όμω όμως χρόνο ότι συμφωνώ απόλυτα με τα όσα μας είπε. Ε, με την αντίδρασή της δηλαδή στη δικιά μου γνωμοδότηση, γιατί αναφέρθηκε στην πολιτική διάσταση της στρατηγικής 2020 και ότι για να πετύχουμε τους στόχους της στρατηγικής αυτής Πράγματι, πρέπει να έχουμε μια πολιτική απασχόλησης πιο προθυμένη. Συμφωνούμε απόλυτα πάνω σε αυτό. Και πιστεύω ότι η δικιά της η προσέγγιση είναι ακριβώς ίδια με τη δικιά μου. Τη στηρίζω λοιπόν απόλυτα. Δεύτερον, θέλω να σας πω ότι χρειαζόμαστε μια θεσμική προσέγγιση που να έχουμε σκεφτεί καλά να σκεφτούμε καλά τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί μόνο τότε προσφέρουμε και νομιμότητα στην πρόταση αυτή. Ίσως όμως, στα πλαίσια των τροπολογιών, να αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε περισσότερο πάνω στο θέμα της νομιμότητας. Προς το παρόν, λέω μόνο ότι δεν είναι αναγκαία η θεσμική προσέγγιση εκείνη που θα λύσει και τα ζητήματα οικονομικής πολιτικής. Απ' την άλλη όμως είμαι πεπισμένος ότι οι τοπικοί φορείς πρέπει να είναι παρόντες, χωρίς όμως να τους επιβάλλεται επιπλέον ε, βάρος σε σχέση με τις στατιστικές για την απασχόληση. Τρίτη μου παρατήρηση. Πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να εκφράσουμε την άποψή μας γνωρίζοντας πολύ καλά ε, τα αποτελέσματα της έρευνας για την ανάπτυξη και προτείνοντας νέες λύσεις υπέρ της απασχόλησης. Αυτό σε συνεργασία με τη συνάδελφο. Τότε πιστεύω ότι θα πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως... Ρότχουλτ, μήπως ε, θέλετε να μιλήσετε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που μας προσκαλέσατε εδώ. Τα διευθυντικά ταμεία γενικότερα, δηλαδή όσον αφορά την παρακολούθηση της στρατηγικής 2020. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό και με το, την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, αλλά και σε αυτές τις διαπραγματεύσεις παρακολουθούμε πολύ καλά τα αποτελέσματα της στρατηγικής αυτής και τις προτεραιότητες. Όπως ανέφεραν και οι ευρωβουλευτές, πρέπει να δούμε πώς θα ενισχύσουμε την απασχόληση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να παρουσιάσει ένα τέτοιο πακέτο και σχεδιάζουμε επίσης να στηρίξουμε περισσότερο το πλαίσιο αυτό ώστε να αλλάξει η κατάσταση όσον αφορά τη μακροχρόνια ανεργία. Για τη συγχρηματοδότηση θέλουμε να ενισχύσουμε την συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους επίσης και άλλους εταίρους μας. Εννοείται ότι προσβλέπουμε και σε ενισχυμένη συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Κανένας άλλος δεν βλέπω να θέλει το λόγο για αυτό το σημείο. Οπότε προτείνω προθεσμία για υποβολή τροπολογιών, η ίδια όπως και για την έκθεση του Τομάς ε, Τότς, 4 Δεκεμβρίου δηλαδή, στις 12 το μεσημέρι. Συνεπώς λύγει το σημείο αυτό. Δεν περιμέναμε να προχωρήσουμε τόσο γρήγορα με την ψηφοφορία, οπότε τελειώνουμε εδώ για το πρωί και θα τα ξαναπούμε στις 4. Όμως στις 2.30 στην αίθουσα Γιάννη 2Q2 υπάρχει μια ανοιχτή συνεδρίαση με τον κύριο Φανερομπάου της διάσκεψης των Πρόεδρων, έτσι για τη διάσκεψη κορυφής, οπότε αν θέλετε μπορείτε να πάτε. Μπορεί να είναι ενδιαφέρον για εσάς που ασχολείστε με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και την πορεία μας προς αυτό. Γι' αυτό και αναβάλαμε την απογευματινή συνεδρίαση, γιατί δεν επιτρέπεται καμία συνεδρίαση συγχρόνως με εκείνη τη διάσκεψη του Πρόεδρου. Παρόλο που δεν θα μπορούμε όλοι να παρευρεθούμε εκεί, γιατί η αίθουσα δεν είναι και τόσο μεγάλη. Εν πάση περιπτώσει, εδώ στις 4 θα τα ξαναπούμε. Και όσοι θέλουν να πάνε στην αίθουσα Γιάννα 2Q2, αρχίζει στις 2.30 και είναι με τον κύριο Φανουρομπάου για την τελευταία διάσκεψη κορυφής. Σας ευχαριστώ, θα τα πούμε το απόγευμα.